εξόπιση ανδρών και γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιριών. Πρώτα θα μιλήσουν οι δύο συντάκτες. Η πρώτη, κυρία Ρέγνερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να μπορούν να εκπροσωπούνται άνδρες και γυναίκες με ισότιμο τρόπο στα διοικητικά συμβούλια, χρειαζόμαστε δεσμευτικού κανόνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διότι από μόνη του κανένα θα κάνει τίποτα. Κανείς. Μόνο στις χώρες εκείνες όπου υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες βλέπουμε να γίνονται πραγματικά βήματα προόδου και να αυξάνονται οι αριθμοί των γυναικών. Δεν μπορεί πλέον να αρκεστεί κανείς σε υπομονή. Το Κοινοβούλιο έκανε τη δουλειά του. Και τι θέλουμε ακριβώς. Θέλουμε στις εισηγμένες σε χρηματιστήρια επιχειρήσεις να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών στο 40% στη βάση αντικειμενικών διαδικασιών. Αντικειμενικών επιμένω. Δηλαδή η βέλτιστη των ανδρών και οι βέλτιστη των γυναικών πρέπει να επιλέγονται. Αυτό θα ωφελήσει και την οικονομία και βεβαίως είναι και αίτημα δικαιοσύνης και περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για πραγματική προσφορά προς τις χώρες μέλη. Υπάρχει στο κείμενο και μια παράγραφο που επιτρέπει σε χώρε όπω η Γερμανία Σε ό,τι αφορά τι εθνικέ προσπάθειε που έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια και που καταβάλουν ακόμη, δηλαδή για να αυξήσουν το ποσοστό των γυναικών στις επιχειρήσεις, αυτά να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή πρόκειται μια, μια πραγματική προσφορά προ τι χώρε μέλη για να δείξουν αυτέ θάρρο και να δεχθούν τα όσα λέει η έκθεση. Ο φάκελος, η επεξεργασία του φακέλου έχει ολοκληρωθεί είναι, έχει τεθεί πλέον επιτάπητος. Γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα την Λουξεμβουργική Προεδρία που δείχνει αυτή την ενέργεια ή καλύτερα την ενεργητικότητα να κάνει μια προσπάθεια, δεν θέλω να πω μια τελευταία προσπάθεια, να κάνει μια προσπάθεια να πείσει και τις χώρες που ακόμα διστάζουν. Πολύ σύντομα, στις 7 Δεκεμβρίου τελείται το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Απασχολήσεως. Απευθύνω έκκληση προς όλες τις χώρες εξετάστε το, τον φάκελο. Ο φάκελος είναι πολύ ήπια, δηλαδή το θέμα μας, ε, το κείμενό μας είναι ήπια διατυπωμένο. Οφελεί και άνδρες και γυναίκες και την ίδια την οικονομία. Και ιδίω εν ώψη του ιστορικού, του δράματος δηλαδή των προσφύγων, πρόκειται για ευρωπαϊκές αξίες που τονίζονται για άλλη μια φορά. Ακόμα λοιπόν πιο σημαντικό είναι να τεθεί και το ζήτημα της ισότητας των φύλων αλλά και της λεγόμενης στα αγγλικά corporate governance. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέγνερ και κυρία Κάπριλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω εσάς κυρία Επίτροπε αλλά και την Προεδρία του Λουξεμβούργου και κυρίως την κυρία Υπουργό, την κυρία Μίτς για τις προσπάθειες που έκανα να προχωρήσει το θέμα όσον αφορά το σχέδιο οδηγίας. Δυστυχώς Δύο χρόνια μετά, η ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, μετά από αυτή την ψήφο, μπορώ να επαναλάβω την ομιλία που έκανα αυτολεξή στην Ολομέλεια τότε. Έκανε τη δουλειά το Κοινοβούλιο και να και στα κράτη-μέλη να ανασκουμποθούν και να εφαρμόσουν τι αναληφθήσει υποχρεώσει για τι ισότητε ανδρών και στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου εν πρώτη να υπενθυμίσω τα γεγονότα, διότι φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν κάποιοι διστακτικοί ε, αμετανόητοι στην οδηγία. Δηλαδή έδειξαν τα γεγονότα ότι η μεγαλύτερη παρουσία στα διοικητικά συμβούλια των γυναικών οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση, καλύτερη κυβέρνηση και καλύτερε οικονομικέ επιδόσει. Τι περιμένουμε λοιπόν ακόμα να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητε των γυναικών και να έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μα για να πετύχουμε του στόχου οικονομικού και κοινωνικού. Δείχνουν επίση τα γεγονότα ότι λειτουργεί η διοικητική πίεση στα πλαίσια της προτάσεως οδηγίας ξέρουν περάσαμε από το 15,8% σε πάνω από 6% των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Ή βλέπουμε ότι έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό αύξηση από τη στιγμή που υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθετική πίεση. Οι επιχειρήσει προβλέπουν, αν θέλετε, προδικάζουν τα αποτελέσματα τη οδηγία και προσλαμβάνουν ικανέ γυναίκε. Θέλω να επιμείνω εκ νέου και στο φαινόμενο χιονοστιβάδα που μπορούμε να περιμένουμε από την οδηγία, θετικά αποτελέσματα σε διάφορα επίπεδα ιεραρχικά, όχι μόνο χάρη στα διάφορα μέτρα που θα εφαρμοστούν. Για εκείνου που δεν έχουν πιστεί, τουλάχιστον να στείστε πραγματιστέ. Δεύτερο σχόλιο γενική φύσεω. Η νομική βάση που επελέγει, τα εργαλεία που επελέγησαν, δηλαδή η οδηγία και η πρόταση που διατυπώθηκε από το Κοινοβούλιο, προσφέρουν ήδη ένα μεγάλο περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη το μόνο πράγμα που περιμένουμε εδώ και δύο χρόνια τελικά είναι μια δέσμευση από πλευρά των κρατών μελών και συγκεκριμένε δράσει, ώστε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Εν κατακλείδη, να πω τρία πράγματα. Ευθύνη χρειάζεται, ευελιξία και συγκεκριμένε προσπάθειε. Και πίσω από κάθε λέξη από αυτέ κρύβονται τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Γκάμπριελ. Κύριε Σμιτ, εξ ονόματο του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Ρέγνερ και κυρία Γκάμπριελ, Καταρχάς να σας συγχαρώ για τη δυνατότητα που μου προσφεράτε ώστε να μπορέσω να μιλήσω στο Κοινοβούλιο και να σας ενημερώσω για το πού βρίσκονται οι εργασίες σχετικές με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόταση οδηγίας όσον αφορά τη βελτίωση της οροπίας ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Όσον αφορά το θέμα αυτό, το Κοινοβούλιο ήδη υιοθέτησε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως ήδη υπενθυμίσατε και εντός αυτής της θέσεως υποστηρίζει ευρέως την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα στοιχεία όσον αφορά την ισορροπία ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 1 πέμπτο των μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες. Είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός, γελία χαμηλός, αλλά δείχνει κάποια πρόοδο. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ υπομονετικοί, ούτω ώστε τελικά να καταλήξουμε με αυτού τους ρυθμού σε ισότητα ή σε ισορροπία. Λοιπόν, υπάρχει ανάγκη, πραγματική ανάγκη να διευθετηθεί αυτό διαφορετικά και να επιταχυνθεί κάπως ο ρυθμός. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το 2010 όταν αυτές οι συζητήσεις ξεκίνησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ένα μέλος στα 10 των διοικητικών συμβουλίων ήταν γυναίκα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την επίθεσή μας κατά του προβλήματος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τον 21ο αιώνα στο Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε κυριαρχία των ανδρών μεγαλύτερη ισότητα στις διευθυντικές θέσεις είναι ένα θετικό μήνυμα που απευθύνεται προς την κοινωνία στο σύνολό της. Η ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών εντός των οργάνων λήψης αποφάσεως είναι σίγουρα θέμα συγκεκριμένο ισότητας, είναι επίσης ένα σύμβολο, αλλά θα προσέθετα ότι αποκαλύπτεται τελικά η ποικιλομορφία αυτή, όπως είπατε κυρία Γκάμπριλ, αποσύρεται πολύ συχνά να είναι θετική από την άποψη της σωστής διακυβέρνησης, χρηστής διακυβερνήσεως των επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, η Προεδρία του Λουξεμβούργου αυτό το θέμα το έθεσε ως μία από τις προτεραιότητές του, τις μεγαλύτερες. Παρουσιάσαμε πολλές νέες προτάσεις συντακτικής φύσεως, ούτως ώστε να εξευρεθεί ένα συμβιβασμό στο Συμβούλιο εντός των φορέων του Συμβουλίου η πρόταση σε αυτή εξετάστηκε ενδελεχώς και συνεζητήθη δόντους Και τώρα, μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις, έχουμε θέσει το σημείο αυτό στο, στην διάταξη του Συμβουλίου Ευσκόπου που θα συνεδριάσει την επόμενη Δευτέρα, ούτω ώστε να υπάρξει ενημέρωση επί του θέματος και να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια ειδική πλειοψηφία α, ε, υπέρ της προθήσεως του ζητήματος. Δεν θα ήθελα να προδικάσω τώρα την διέξοδο, το αποτέλεσμα των συζητήσεων εντός του Συμβουλίου, αλλά μπορώ δυστυχώς να σας ανακοινώσω ήδη ότι οι πρόσφατες συζητήσεις στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές. Σήμερα είχα πολύ καλή είδηση που άκουσα διότι έμαθα ότι μια χώρα που γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Επίτροπε, πράγματι ανακοίνωσε ότι άλλαξε θέση. Δηλαδή απαρνητική θέση εκινήθη προς Και αυτό πιστεύω είναι ένα καλό μήνυμα, είναι ένα σημάδι άκρος θετικών. Όπως γνωρίζετε, αυτή η πρόταση εμπεριέχει διαδικαστικούς κανόνες περιοριστικής φύσεως που στοχεύουν την επίτευξη των ποσοτικών στόχων. Απαιτείται η διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ακριβοδίκαια, εδραζομένη επί των προσόντων και της διαφανείας. Οι βασικές δυσκολίες απορρέουν από το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη ή τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις Κάποια κράτη-μέλη είναι σε πιο προθυμένο στάδιο από ό,τι άλλα όσον αφορά το βαθμό ισότητας ανδρών γυναικών στο επίπεδο αυτό που συζητούμε. Εν γέννη, θα έλεγα ότι υπάρχει συνένεση υπέρ του στόχου της προτάσεως. Αλλά αν ο μεγάλος αριθμός των κρατών μελών δηλώνει ότι είναι θετικό για μια νομοθεσία σε επίπεδο ένωσης, άλλες χώρες και δυστυχώς για την ώρα ακόμα αποτελούν μια μειονότητα που μπλοκάρει το θέμα. Υπάρχει διαφορά, υπάρχουν διαφορές σε εθνικό επίπεδο. Προωθούν το θέμα της επικουρικότητας, προωθώντας εθνικές ιδιαιτερότητες ή συστήνουν μη περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες που δημιουργούνται να στέλνουν μια ψηφία. Η Προεδρία επεξεργάστηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για ισότητα ανδρών και γυναικών ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία υιοθετούνται και θα υιοθετηθούν, πιστεύω τα καταφέρουμε, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ της 7ης ε, Δεκεμβρίου. Βασίζεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα ανδρών και γυναικών, ε, που αναφερόταν στην όλη παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη, Πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να ωφεληθούν από τα ταλέντα και τον δυναμισμό και των ανδρών και των γυναικών. Η Ευρώπη διαθέτει πάρα πολλά ταλέντα ανεκμετάλλευτα και πάνω απ' όλα σήμερα βλέπουμε ότι 60% των διπλωματούχων με πτυχίο πανεπιστημιακό στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Συνεπώς δεν υπάρχει ουδής λόγος τον 21ο αιώνα οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες ή οι άλλοι θεσμοί ακόμα βασικά να διευθύνονται από άντρες. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διατήρησε το θέμα της ότης ανδρών και γυναικών στην ημερήσια διάταξη και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα εμπνεύσει στη συνεδριά του Συμβουλίου ε, τα μέλη του Συμβουλίου στη συζήτηση που διεξαχθούν στις 7 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ Σμίτση. Και τη συζήτηση την ξεκινάμε με την κυρία Λεγκρίπ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, απόψε δεν είμαστε πολλοί εδώ μετά από την ε, ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση της έκθεσης ε, Ρέγνερ για να μιλήσουμε για μια ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών ε, σε, σε επίπεδο λήψη αποφάσεων, στα όργανα λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των γυναικών. Έχουμε ένα καλό και ένα κακό νέο από ό,τι μας είπατε κύριε Υπουργέ Συμφωνούμε μαζί σας και με την Επίτροπο θεωρούμε ότι επιτελείται πρόοδος και το είδαμε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο Υπουργών, όπως είπε η συνάδελφος όμως Μαρία Γκαμπριέλ, από πλευράς ε, Ευρωκοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση υπάρχει μια διαφάνεια, μια δέσμευση και μία πραγματιστική προσέγγιση για να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας, την θέση των κρατών μελών και τις επιθυμίες τους. Έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, έχουμε κάνει βήματα προς τα μπρος, χωρίς να απαρνηθούμε τις δεσμεύσεις μας για μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι μπορούμε να μιλάμε για ποσοστώσεις γιατί στη Γαλλία ε, υπάρχει ένας νόμος από το 2011 ο οποίος ε, έδωσε αποτελέσματα. 33 δηλαδή της 100 συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων. Θεωρούμε όμως ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές νομοθετικές προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει, όπως είπαν και άλλοι, να λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διασπαθίζουμε το ταλέντο των γυναικών που έχουν μια πολύ υψηλή κατάρτιση. Και αυτό έχει σημασία για τις γυναίκες και για τα παιδιά. Ευχαριστούμε κυρία συνάδελφε Λεγκρίπ. Για ένα, ένα μισή λεπτό η κυρία Χέκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Στι 14 Ιουλίου 2015 η Προεδρία από πλευράς Λουξεμβούργου τοποθετήθηκε θετικά όσον αφορά την οδηγία για τις ε, ανώτερες ε, θέσεις ε, στις επιχειρήσεις για τις γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σα βλέπουν σημαντική ανάγκη να υπάρξει μια οδηγία. Μεγαλύτερη ισότητα στις ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων οικονομικά και με επιχειρήματα υπέρ των γυναικών να προωθείται βασίζεται ω ότι οι επιχειρήσεις θα κερδίσουν αν έχουν περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Έχει λοιπόν και οικονομικούς λόγους και είναι επιτέλους η χρονική στιγμή που ήρθε μετά από πολλά χρόνια τα πατριαρχικά δίκτυα να αποσυναρμολογηθούν, να διαλυθούν σε σχέση με τις ανώτερες ε, ηγετικέ θέσει. Μέχρι σήμερα είχαν οι άνδρες καλύτερε θέσει, τώρα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Στην συνέχεια η κυρία Φωνστόχη παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο με κάθε τρόπο θέλει να περάσει ποσοστό υπέρ γυναικών. Είναι απόλυτα λάθος αυτό. Γιατί, γιατί ποσοστώσεις για ηγετικές θέσεις αν δεν υπάρχουν είσαι και για την πυροσβεστική ή για μηχανολόγους και μηχανικούς και γιατί μόνο για γυναίκες και όχι και για τους αμφιφιλικούς και τους διαφιλικούς. Και βλέπουμε εδώ ότι όταν έχουμε μονομερή τέτοια ε, κατάσταση, έχει την ελευθερία μια επιχείρηση να προσλάβει γυναίκες ή άνδρες ε, όσους επιθυμεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια με διαφορά σε σχέση με τις διακριτικές, μετα... τη διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλλο και αυτό απορρίπτουμε φυσικά όπως και τις ποσοστώσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φωνστόχ. Κυρία Φωνστόφια, επιτρέπετε μία ερώτηση από πλευράς Ρέγνερ, συναδέλφου Ρέγνερ. Παρακαλώ συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Μα ακούτε τώρα, εντάξει. Την έκθεση τη διαβάσατε. Στην έκθεση αναφέρονται διαδικασίες, δηλαδή αντικειμενικές διαδικασίες, ο στόχος. Και δεν αναφέρεται στην έκθεση ότι πρόκειται για ποσοστώσεις. Το διαβάσατε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ο στόχος είναι ποσόστοση 40% στα διοικητικά συμβούλια. Αυτή είναι η αρχή, η έναρξη και είναι λάθος. Ο στόχος είναι μια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών, διότι θα προσλαμβάνονται ως γυναίκες και χωρίς άλλα προτερήματα ή προσόντα. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο εμείς ε, απορρίπτουμε. Σας ευχαριστούμε, λέγει Πρόεδρος. Στη συνέχεια η κυρία Μπιμπάου Μπαραντίκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα στην Ευρώπη 6 από κάθε 10 φοιτητές είναι γυναίκες Ωστόσο, 8 από κάθε 10 συμβούλους στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι άντρες. Αυτό είναι ανισότητα, άδικο, κοστίζει χρήματα εις βάρος μας και είναι εις βάρος της Ένωσης. Και πρέπει να επιληθεί αυτό. Οι ποσοστώσεις έδειξαν ότι είναι αποτελεσματικές για να επανορθωθούν τέτοια προβλήματα. Αρκεί μια πολιτική απόφαση που θα διευκολύνει την πρόσληψη γυναικών στις ηγετικές θέσεις επιχειρήσεις και θα διευκολυνθεί και η ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν Όπω όπως σε σχέση με το όσα ότι οι επιχειρήσεις που έχουν περισσότερη ισορροπημένη σχέση γυναικών είναι πιο ανταγωνιστικές. Έχουν καλύτερο τζίρο και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λειτουργούν καλύτερα και δημιουργούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πελάτες και στους επενδυτές. Γι' αυτό πρέπει να εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα στρατηγικά και με καινοτόμο τρόπο. Πρέπει να ξεκινήσουμε με δημόσια προγράμματα ώστε να ξεκινήσουμε να επιτυγχάνουμε επενδύσεις. Είναι λοιπόν αυτό προτέρημα επενδυτικό για να γίνει γίνουμε πρωτοπόροι παγκόσμια. Διαφάνεια και ισότητα στην επιλογή λοιπόν των ατόμων που θα συναπαρτίζουν ε, το Διοικητικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε από πλευρά τη Επιτροπή ε, για την προσπάθεια που γίνεται να προαχθεί αυτή, ε, αυτός ο στόχος. Να αναθεωρήσουν οι χώρες τις θέσεις τους και να κατανοήσουν ότι ενώ υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις τα μεγάλα προγράμματα για ισότητα θα είναι χαρτί το οποίο δεν θα αξίζει καθόλου πια. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ακολουθεί η κυρία Φορέτσα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λυπάμαι γιατί άκουσα μία συνάδελφο να αγνοεί ένα ζήτημα γιατί από τις 5 Νοεμβρίου οι γυναίκες ε, στην ουσία εργάζονται με βάση αυτό το χάσμα αμοιβών ανδρών-γυναικών. Άρα δεν μιλάμε για ποσοστώσεις για να προωθήσουμε τις γυναίκες. Θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερες διακρίσεις σε σχέση με τις γυναίκες, γιατί οι διακρίσεις είναι πολύ υψηλές στα διοικητικά συμβούλια και όχι μόνον. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ποιες είναι οι στρατηγικές για να καταρρίψουμε αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε οι άνδρες και οι γυναίκες να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό η κυρία Ράιντκε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπη, κύριε Σμίτ. Θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά απλό. Έχουμε ένα κοινό πολιτικό στόχο, ισότητα δηλαδή γυναικών και ανδρών. Εδώ σε σχέση με τις ηγετικές θέσεις επιχειρήσεις έχουμε εργαλεία και μέσα που λειτουργούν, δεσμευτικοί κανόνες για τους οποίους έκανε λόγος η συνάδελφος και όλοι θα υποφελούμεθα, γυναίκες και άνδρες από αυτό στην κοινωνία μας. Η πολιτική μπορεί να είναι καμιά φορά τόσο απλή υπόθεση. Όμω σε κάποια κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Κυρίω η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τη Γερμανία. Και αυτή τη στιγμή αγαπητή κυβέρνηση τη Ομοσπονδιακή Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο αίτημα. Τώρα να μην εγκρίνεται αυτή την πρόταση, όχι μόνο λάθο, θα ήταν και παράλογο και η Υπουργό Οικογενειών στη Γερμανία που υποστηρίζει αυτή την πρόταση να γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο σας υποστηρίζει. Να ξέρετε ότι η πρόταση την επόμενη Δευτέρα μπορεί να επιτύχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο με την ψήφο της Γερμανίας. Ευχαριστούμε συνάδελφε Ράινκε. Για 1,5 λεπτό η συνάδελφος James παρακαλώ. Κοιτάξτε, η συνεισφορά μου σημερινή συζήτηση θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία μου που ήμουνα πρώην μην, α, ήμουν στο χρηματιστήριο, σε μια εταιρεία του χρηματιστηρίου, σε καταπίστευμα. Και μετά ήμουν επίσης και μέλος άλλων φορέων. Λοιπόν, δεν λαμβάνει υπόψη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι κάτι που είναι ενδυμικό στην κοινότητα την επιχειρηματική. Δεν είναι αυτό που ξέρεις, αλλά ποιον ξέρεις που παίζει ρόλο. Ακόμα και στο διεθνή τομέα για προσλήψεις που είναι υπεύθυνοι για το κυνήγι κεφαλών και προσόντων βλέπουν ότι είναι αυτή η υποκαδιατική κατάσταση που κρατεί. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες να έχουν ε, ρόλο επιρροή στις επιχειρήσεις, να στο διοικητικό συμβούλιο. Τελικά η πραγματικότητα στρέφεται κατά αυτού. Το διακύβευμα δεν αφορά την εμπειρία, τα προσόντα και τα ταλέντα τους, αλλά τη διαφάνεια όσον αφορά τις προσλήψεις και τη συνεισφορά τη ποιοτική προσλήψεω. Η ποιοτική πρόσληψη είναι όπως κάτι διαφορά. Δεν έχει σχέση το φύλλο και μέσω της αγωγής ε, ποσοστώσεων η καταπολέμηση της διακρίσεως τελικά καταπνίγεται από τη διάκριση. Θα πρέπει να έχουν ποσοστό 40% οι εταιρείε, θα έχουν κυρώσει εάν δεν το κάνουν και αυτό δεν είναι υπεύθυνο ούτε ρεαλιστικό σαν νομοθεσία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να λύσει το πρόβλημα Πηγαίνετε πίσω ξανά στο σχεδιαστήριο και αντιμετωπίστε ε, το κατεστημένο που είναι γεμάτο από εκείνους που μισούν τις γυναίκες και δημιουργούν ένα δίκτυο που στηρίζει τους άντρες στην Ευρώπη. Δεν μπορώ όμως να στηρίξω αυτό το μέτρο. Ευχαριστούμε συνάδελφε Τζέμις. Για ένα λεπτό Μπονάνο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα σε σχέση με μια σύγκριση που θέλω να κάνω όσον αφορά τις ε, γυναίκες στις χώρες, ακόμα και στην Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει μια μέθοδος για τις γίνεται γενετικός ακοτηριασμός στα μικρά κορίτσια. Λοιπόν, αυτά γίνονται σε χώρες τις μουσουλμανικές και μετά έρχονται οι μουσουλμάνες στην Ευρώπη και γίνονται στα μικρά κοριτσάκια μόνο για λόγους ε, θρησκευτικούς. Και εμείς μιλάτε για τις γυναίκες, τις εταιρείε, για τις γυναίκες που πρέπει να είναι παντού, αλλά δεν καταπολεμείτε αυτό, αυτή την ασκήμια εκείνων των ζώων των κτηνοδιών που κάνουν στα κοριτσάκια, στα μωρά. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση των γυναικών. Μόνο για τα διοικητικά συμβουλίου σας ενδιαφέρουν μόνο τα χρήματα και θέλετε να, να παριστάνουν μονάχα ε, σαν μοντέλα στη μόδα. Και αυτή την κτηνοδία της γενετικής ακροτηρίασης που σαν κτίνοι οι μουσουλμάνες ε, βλάπτουν διαβίου αυτές τα, αυτά τα κοριτσάκια όταν γίνουν γυναίκες. Αυτό είναι μια πραγματική ασκήμια. Σε ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Βουναν, Επιτρέπετε μία ερώτηση από την κυρία Μπιλμπάο, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο κυρία Μπιλμπάο, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι όλοι μας συζητήσαμε εδώ σχετικά με αυτό το θέμα και θα σας παρακαλούσα και εσείς να προσαρμόζετε, προσαρμόζετε σε αυτό. Δεύτερο, θα σας παρακαλούσα να είσαστε παρόν σε όλες τις συζητήσεις που έγιναν σε αυτό το σώμα για την ισότητα, τη διακριτική μεταχείριση και τα δεινά που υφίστανται πολλές γυναίκες στον κόσμο και τα κορίτσια και οι γυναίκες από άλλες περιοχές και υπήρους. Και αναφέρομαι ε, στον γενετικό ε, ακροτηριασμό. Δεν είσαστε όμως σε αυτές τις συζητήσεις και θα ήθελα, διακόπτεται η ομιλήτρια. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου Μπαράντικα. Κυρία συνάδελφε, κατανοώ φυσικά το ότι ζητείτε να παρέμβετε αλλά λυπούμε. Δεν ήταν ερώτηση φυσικά που, αυτό που διατυπώσατε στον συνάδελφο. Ο κύριος Μπονάνο. Να υπογραμμίσω ότι είμαστε, είμαι σε 22-22 αυτή θέση σαν παρουσία σε σειρά των βουλευτών, σαν δουλειά που κάνω. Λοιπόν, δεν μου θα μου κάνετε εσείς μαθήματα. Μπα κάνω εγώ μαθήματα σε εσά. Εγώ μιλάω για εκείνο που συμβαίνει στον κόσμο με τις γυναίκες. Εσεί μιλάτε για διοικητικά συμβούλια. Αλλά ντραπείτε Εσεί είσαστε μόνο αριβιστέ, σκεφτόσαστε μόνο την εξουσία, δεν σκεφτόσαστε τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, στι γυναίκε. Ε, ε, ε, είσαστε σικ κομμουνιστέ και τρώτε χαβιάρι και σαμπάνια και γεμίζετε το στόμα σα. Αυτό είσαστε εσεί. Σε ευχαριστούμε συνάδελφε Μπονάνο. Συνάδελφε Μπονάνο. Η συζήτηση για αυτό το θέμα έγινε επί του οποίου αναφέρθηκε η συνάδελφος. Η συνάδελφος Σουίτσα παρακαλώ έχει τον λόγο. No, no, no, Όχι, δεν γίνεται αυτό. Συνάδελφε Σουίτσα, έχετε τον λόγο. Συνάδελφος Σουίτσα έχει τον λόγο. Ε, λοιπόν, κύριε Μπονάνο, διέκοψε την ιδηλιακή συζήτηση εγώ θα προτιμούσα να συμμετείχαν περισσότεροι άντρε στη συζήτηση, να μην είναι μόνε οι γυναίκε που το κουβεντιάζουν. Φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και προσπαθούμε να περάσουμε τη θέση μα. Δυστυχώ πρέπει να πω ότι όσο μεγαλώνω, τόσο είμαι υπέρ των ποσοστώσεων. Η κοινωνία απλώς δεν θα γίνει δίκαιη μέχρι τη στιγμή που οι γυναίκες εκπροσωπούνται εξίσου. Μέχρι να έχουμε 50-50% συμμετοχή των γυναικών ή πάνω από 50%. Βέβαια με τις ίσες δυνατότητες και τις δίκες διαδικασίες όπως ήδη ε, αναφέρθηκε. Έχουμε τεράστια πρόοδο εν συγκρίση με το 2010. Αυτό το είπε ο κύριο Σμιτ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Λουξεμβούργου που έχει δώσει ύψη τη σημασία στο θέμα, διότι από 11% φτάσαμε στο 21% εκπροσωπήσεω των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πιστεύω ότι αυτή είναι πρόοδο, αλλά όχι επαρκή. Μα είπατε να είμαστε υπομονετικοί. Οι γυναίκε είναι φημισμένε για την υπομονή του, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι και η ώρα η ισότητα των φύλων να επιτευχθεί και να φαίνεται και στα διοικητικά συμβούλια. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Τα κράτη-μέλη όμως είναι εκείνα που θα πρέπει να αντιδράσουν και τη Δευτέρα, 7η Δεκεμβρίου, περιμένουμε να ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν αυτές τις χώρες και τελικά να δεχτούν οι χώρες που δεν, που δέχτηκαν μέχρι τώρα την οδηγία. Εκεί που υπάρχει αναγκαία νομοθεσία είναι προφανές ότι ο κόσμος συμπεριφέρεται διαφορετικά στις χώρες αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω και να σας ζητήσω εφόσον το Κοινοβούλιο έκανε τη δουλειά του, να συνεχίσετε τις προσπάθειες και στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τις πτυχιούχους γυναίκες που είναι 60% του πληθυσμού εν συγκρίση με τις, με, μάλλον 60% γυναίκες πτυχιούχες εν συγκρίση με 66% άντρες. Ε, λοιπόν είναι σαφές ότι σε όλες τις χώρες δεν μπορούμε να, έχουμε, ε, να δεχτούμε την κατάσταση που επικρατεί στη Μάλτα Υπάρχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χάνιμπολ, παρακαλώ. Μικρό. Ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Λουξεμβουργιανή Προεδρία για το καλό της έργο σε αυτό το θέμα. Το επανέγραψαν στην ημερησία διάταξη. Δεν έπρεπε ποτέ όμως να έχει εγκαταλείψει αυτή την ημερησία διάταξη. Όπως πολλοί προανέφεραν, προλαλήσαντες, χώρες με περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια έχουν καλύτερες επιδόσεις από ότι τα διοικητικά συμβούλια μόνο με άνδρες. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει το ορθό αυτή τη θέσεω. Όμω δεν έχουμε φτάσει στην ισότητα ακόμα. Πόρο απέχουμε. Και σαν αποτέλεσμα φυσικά χάνουμε ε, μεγάλα ταλέντα τα οποία χάνονται ενώ από πλευρά των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια υπάρχει αύξηση, δεν είναι αρκετή αυτή η αύξηση. Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε και σε σχέση με το 25% των μη εκτελεστικών διοικητών είναι γυναίκες και στο Ηνωμένο Βασίλειο η συντηρητική κυβέρνηση αποτελεί τμήμα της τροχοπεδούσας μειονότητας συγκεκριμένα ανέφερα μη εκτελεστικές θέσεις ε, διευθυντών, διότι αυτό είναι το θέμα της έκθεσης. Και πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Πρέπει να υπάρξουν εκτελεστικοί διοικητές ε, γυναίκες. Ε, ευχαριστούμε κυρία Χανιμπορ. Για ένα λεπτό η κυρία Ζιτνιάνσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Απόψε δεν είναι το θέμα αν είναι καλό ή όχι να έχουμε περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, αλλά είναι καλύτερο οπωσδήποτε να μπορεί να υπάρχει πολυμορφία και να την πετύχουμε. Αυτό και σε σχέση με τις εθνικές και εθνοτικές διαφορές θα έπρεπε να ισχύει και για τα άτομα με ιδιαιτερότητες ή ειδικέ ανάγκες θα μπορούσαν με ποσοστώσεις να προχωρήσουν ε, οι προσλήψεις αυτών των ατόμων. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει πολλά επιχειρήματα υπέρ αυτού στην κοινωνία μας. <clears throat> Δεν νομίζω ότι είναι όμως ε, αναγκαίο από την άλλη πλευρά σε όλες τις χώρες. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες ε, να προαχθούν ε, αν ε, δεν γίνεται με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία και μέσα σε σχέση με τη συνεργασία με τους άντρες για τις υποδομές στις οικογένειες από πλευράς πολιτικής και πολιτικά υπεύθυνων θα πρέπει να προαγάγουμε διαφορές και αναδιαρθρώσεις ώστε να προχωρήσουν οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζητνιάσκα. Η κυρία Βίξτρομ δεν παρίσταται. Για ένα λεπτό η κυρία Γιούτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι από το κίνημα των πέντε αστέρων, είμαστε κατά αυτή τη τάση, είτε πρόκειται για το χρηματιστήριο είτε για την πολιτική. Γιατί η πραγματική συμμετοχή των γυναικών θα πρέπει να είναι καρπός των δικών μας ε, ικανοτήτων και να ορίζονται αξιοκρατικά διαφανή κριτήρια με ισότητα για όλους. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει μία διευθυντική θέση να αναθέτεται σε γυναίκα επειδή είναι γυναίκα. Θεωρούμε όμως ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη αξία. Ελαμβάνουμε υπόψη αυτή την ελληματική διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως ίσχυσε και με την οδηγία για την μητρότητα. Δυστυχώς το Κοινοβούλιο δεν αντέδρασε στο Συμβούλιο. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν σαφείς αποφάσεις και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι απαράδεκτη η στάση που κρατούν. Ευχαριστούμε κυρία Αγιούτο. Για ένα λεπτό η κυρία συνάδελφος Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Σμιτ, κύριε Επίτροπε, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 30% ποσόστοση γυναικών και αυτό μπορεί να θεωρηθεί θετικό. Κάθε τέταρτο στις επιχειρήσεις στη Γερμανία ε, είναι γυναίκα 26,5% οι γερμανικές επιχειρήσεις νομοθετικά υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυτές τις ποσοστώσεις. Για διοικητικά συμβούλια θα ε, συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα το θέμα ώστε να μπορέσουν να προαχθούν οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια στις μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι το 2020 και να φτάσουν το 40% είναι και προβληματική η κατάσταση σε σχέση με τις αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιες ποσοστώσεις. Τουλάχιστον για κάποιες ε, ε, χώρες η αρχή της επικουρικότητας λαμβάνεται υπόψη. Η πολυμορφία σε σχέση με τα φύλλα έχει θετικές επιπτώσεις επιχειρήσεις. Στη Γερμανία βλέπουμε ότι όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό στα συμβούλια των γυναικών υπάρχουν καλές επιδόσεις από αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν το φύλλο, η ισότητα των φύλων πρέπει να προαχθεί. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κάπερ. Τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Σόιντροβα παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, φοβάμαι ότι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά είναι τα θέματα ασφαλείας, σημαντικότατα ζητήματα. Όμως, ναι, έχει σημασία το φύλλο και είναι σημαντικό που ασχολούμεθα και με ζητήματα όπως αυτό. Η τσεχική κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να μπει στη λέσχη των χωρών εκείνων που ακολουθούν θετική προσέγγιση όσον αφορά αυτό που συζητούμε και δήλωσε σαφώς ότι είναι υπέρ μία ισορροπημένης εκπροσωπήσεως των γυναικών στα συμβούλια, αυτό που συζητούμε. Όμως, Θέλουμε οι γυναίκες να εκπροσωπούνται καλώς στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στην τσεχική δημοκρατία έξι εταιρείε θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του μέτρου. Νομίζω ότι δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα άλλα μέσα που είναι στη διάθεσή μας. Και δεν μου αρέσει το γεγονός ότι ξεκινούμε με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τις δημόσιες επιχειρήσεις, από τις κυβερνήσεις μας, από του περιφερειακούς φορείς. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν το θέμα τα ίδια και οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαπιστώσουν ότι είναι προς συμφέρον τους να έχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια τους. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κυρία Αρένα παρακαλώ. Ευχαριστώ τη Λουξεμβριανή ε, Προεδρία και τον κύριο Σμιτ καθώς ε, και την κυρία Μίνσου για την προσπάθεια που έχουν προσδώσει σε αυτό το θέμα. Μιλάμε λοιπόν για ελάχιστη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Μιλάμε για ένα 21% και ήδη προελέχθη ότι σε ορισμένε χώρες έχουμε ένα 30% ενώ σε άλλες χώρες φτάνουμε στο κατώτατο 2,5%. Όταν μιλάμε για νομοθετικές ε, διαδικασίες ε, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διακρίσεις εκεί που δεν υπάρχει νόμος. Εκεί υπάρχει ανισότητα και δεν υπάρχει θέληση συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θέλουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο Ποια ήταν τα επιχειρήματα των κρατών μελών που αντιτάχθηκαν για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους και να βρούμε λύσεις. Εμείς θα θέλαμε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Αρτένα. Για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι ε, συμφωνούμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ε, επίπεδο διεύθυνσης και συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Τα πράγματα όμως βελτιώνονται. Νομίζω ότι ο καλύτερος άνθρωπος ε, για αυτή την εργασία είναι οι γυναίκες. Ε, δυστυχώς όμως υπάρχει μία κακή προσέγγιση. Πιστεύω στην αξιοκρατία αλλά πιστεύω και στην επικουρικότητα και η κυβέρνησή μου έχει προβάλει αντιρρήσεις για λόγους επικουρικότητας. Άρα δεν περίμενα να δω πράγματα που να με ενδιαφέρουν στο Συμβούλιο. Αλλά διάβασα το άρθρο 4 για την ευελιξία. Ευχαριστούμε Λουξεμβούργο. Κάποιος φαίνεται ότι ακούει. Και ίσως έχουμε την απαρχή μια συμφωνίας εδώ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Γκέρλινγκ. Ακολουθεί για 1,5 λεπτό η κυρία κοζουλοφσκα Ραϊεβίτς. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Μιλούσαμε πολλές φορές για αυτή την οδηγία στο Κοινοβούλιο και μιλήσαμε για τα κέρδη που μπορούμε να πετύχουμε από αυτό. Πολλοί φορείς και οργανισμοί θέλουν να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όσον αφορά τους διοικητικούς φορείς, τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε. Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία ε, και Σουηδία ε, ήταν αναστέλουσα μειοψηφία όσον αφορά το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Αυτή αναστέλουσα μειοψηφία σχηματίστηκε για διαφορετικούς λόγους. Έχουμε Δανία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία, χώρες στις, οι οποίες αντιμετωπίζουν το θέμα με μεγαλύτερη ένταση και έχουν πολλές διαφορετικές λύσεις που εφαρμόζουν. Η Γερμανία έχει ποσοστώσεις, η Σουηδία έχει ξοδέψει όλα χρήματα για τα προγράμματά της, αλλά αυτές οι χώρες που νοιάζονται για αυτό το στόχο είναι στη διαφορετική ομάδα από τις χώρες εκείνες που δεν θέλουν να αντιδράσουν και υπάρχουν ε, πολύ λίγες γυναίκες που είναι στα διοικητικά του συμβούλια και δεν θέλουν να αλλάξει την κατάσταση. Άρα θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με διαφορετικό τρόπο με αυτές τις δύο διαφορετικές ομάδες των χωρών. Εκείνου που θέλουν να πετύχουν το στόχο της οδηγίας και εκείνες τις χώρες που δεν θέλουν να πετύχουν τους στόχους της οδηγίας. Ίσως πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικέ μέθοδοι για την επίτευξη του στόχου θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ή να ε, συμφωνηθούν στα πλαίσια τη οδηγία. Τι ο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μα, δηλαδή οι γυναίκε τελικά να σπάσουν αυτή την οροφή, αυτό το όριο, την αόρατη οροφή, ούτω ώστε οι γυναικείες ικανότητες να μην πηγαίνουν χαμένες και να μπορούν να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε κυρία Κοσλός Καραγεύση. Για ένα λεπτό η κυρία Μούντι τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω ευχαριστίες προς την Λουξιμβουλιανή Προεδρία για το έργο της. Είναι εκπληκτικό να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στο έτος 2015 και ακόμα πρέπει να δίνουμε σκληρά μάχες για την ισότητα των φύλων. Παράλληλα με τους συναδέλφους, πολλούς συναδέλφους σήμερα, να σκεφτούμε πώς μπορεί να επιτεθεί και έγινε πρόοδος για την οδηγία και να αντιληφθούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση άμεσα, εδώ και τώρα. Έχουμε απογοητευτεί σοβαρά από τις αποφάσεις ε, να προσαρμοστεί η γονεϊκή άδεια για τις γυναίκες ε, και πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές για το θέμα της ισότητας των, των φύλων και αυτή η οδηγία δεν είναι μόνο για κάποια θέματα διαδικαστικά. Είναι για την αλλαγή του πολιτιστικού και πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Με περισσότερες γυναίκες σε ηγετικέ θέσεις που μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα όχι σε αυτές τις θέσεις μόνο αλλά σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης. Το να βοηθήσουμε να υπάρχουν γυναίκες στην κορυφή μπορεί να βοηθήσει για μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ισότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφε Μούντι. Για ένα λεπτό η κυρία Τόμασιτς παρακαλώ. Ευχαριστώ οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια, στα συμβούλια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Παρότι συζητήσαμε αυτό το πρόβλημα στο σώμα στην Ευρωβουλή πολλές φορές κατά το παρελθόν. Όλοι συμφωνούμε ότι η μια ηγετική θέση στις επιχειρήσεις πρέπει να έχει ίδια ίση προσπελασιμότητα για γυναίκες όπως και για άνδρες. Πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες όπως και οι άνδρες οι γυναίκες γιατί είναι εξίσου να μαθαίνουν και μπορούν να έχουν ηγετικό ρόλο ρόλο ε, ως ηγέτιδες ε, εργαζομένων. Πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο, το αξίζουν οι γυναίκες, με τη σκληρή τους δουλειά και όχι λόγω φιλανθρωπίας. Κάθε γυναίκα που πραγματικά με αγώνα κατέκτησε μια τέτοια υψηλή θέση με τις γνώσεις της και τα προσόντα της, εξυπηρετεί τα μάλιστα, τα μάλα την, το σκοπό μας και, το, και τους στόχους μας. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των Ευρωπαίων πολιτών και να απαγορευτεί κάθε μορφή διακριτικής μεταχείρισης, θετική αρνητική. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Για 1,5 λεπτό, Πετήρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. 400 από τις ε, μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κροατίας έχουν ε, συμμετοχή γυναικών κατά 15% και 21% στις μικρότερες. Μιλάμε για αυτή τη διαφανή οροφή, αλλά δεν έχουμε επιτύχει πρόοδο. Ιδιαίτερα στην άκρη της ε, πυραμίδας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι ίσως οι ποσοστώσεις οδηγήσουν σε καλύτερη εκπροσώπηση των ε, γυναικών. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς ποσοστώσεις. Βέβαια, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει οι γυναίκες να λάβουν συγκεκριμένες θέσεις ακριβώς επειδή ε, είναι γυναίκες. Απλώς να το δούμε και αξιοκρατικά, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες ε, έχουν τα προσόντα. Ο χώρος των επιχειρήσεων δεν μπορεί να μόνο στους άνδρες. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, έχουμε τις προδιαγραφές και θα πρέπει να επιμείνουμε στην εφαρμογή τους. Αλλά να ε, μην προσκρούσουμε στην ε, επικουρικότητα. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφε Πετήρ, συγγνώμη που χτύπησα με το σφυράκι νωρίτερα. Για ένα λεπτό η συνάδελφος Στάινρουκ τώρα παρακαλώ. Από το 2010 αυξάνεται η ποσόστοση των γυναικών στα συμβούλια των επιχειρήσεων στην Ευρώπη Α, σιγά σιγά. Είναι μια μικρή... Ε, ρογμή αυτή που επιτρέπει να προχωρήσουμε αλλά μια μικρή ρογμή ένα μικρό άνοιγμα θα πρέπει όπως ζητήθηκε από την Ευρώπη να μπορέσουν οι γυναίκες να εκπροσωπούνται στα συμβούλια ώστε μέχρι το 2020 να φτάσουν στο ποσοστό του 40% σε αυτά τα συμβούλια οι γυναίκες. Το Κοινοβούλιο από το 2013 έχει συμφωνήσει. Εδώ και δύο χρόνια αναμένουμε να κινητοποιηθεί κάτι στο Συμβούλιο. Οι εθελοντικές συμφωνίες, οι εθελούσες συμφωνίες δεν φέρνουν αποτελέσματα. Είδαμε στις χώρες όπου υπάρχουν δεσμευτικές τέτοιες συμφωνίες κινητοποιήθηκαν με θετικό τρόπο κινήθηκαν τα πράγματα. Δεν κατάλαβε Πώς η δική μου χώρα, μια και υπάρχει ε, δεσμευτική ποσόστοση στα συμβούλια, κάτι κινήθηκε, αλλά υπάρχουν χώρες που είναι εναντίον και πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Γι' αυτό αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος Μαρία Ρένα, πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα. Τίποτα δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Πρέπει να αποτελέσει αυτό μια βάση για όλους τους Ευρωπαίους γυναίκες και άντρες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφε Στάνρου. Για 1,5 λεπτό η συνάδελφος Κομοντίνη Κάκια παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι την απογοήτευση που υπάρχει από, ε, όπως ε, λέχθη από τους άλλους και ισχύει και στη Μάλτα. Θεωρήσαμε ότι θα είχαμε μία φεμινιστική κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς έχει μειωθεί η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγεσία. Το Συμβούλιο θεωρήθηκε ότι η ισότητα των φύλων είναι ύψιστη της σημασίας για τη σωστή εκπροσώπηση των γυναικών, ενώ εδώ, τη στιγμή που μιλάμε για μη εκτελεστικέ θέσει, Φαίνεται ότι δεν υπάρχει υποστήριξη των κρατών μελών. Φαίνεται ότι ακόμα και στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να προωθήσουν το θέμα για την ισότητα των φύλων. Μιλάμε για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών που υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν γυναίκες με προσόντα. Ακόμα και στη Μάλτα ε, εξελέγησαν περισσότερες γυναίκες βουλευτές από ότι άνδρες στο Κοινοβούλιο. Ε, δυστυχώς δεν υπάρχει ίση εκπροσώπηση, θα πρέπει εκπροσώπηση. Τα μη δεσμευτικά μέτρα είναι ανεπαρκή. Δεν θέλουμε βεβαίως να δημιουργήσουμε γραφειοκρατικές δομές, αλλά θα θέλαμε αυτή η δημόσια και κοινωνική ευθύνη να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Ευχαριστούμε συνάδελφε Κομοντίνη Κάκια. Για ένα λεπτό η συνάδελφος Γιονγκέριους. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είπε ότι ο κόσμος ε, κατά το 2095 ελπίζει το φόρουμ ότι θα γνωρίσει ο κόσμος την ισότητα των φύλων, την ισότητα των ευκαιριών θα θέλαμε να μην περιμένουμε μέχρι τότε για να επιτευχθεί αυτό. Τουλάχιστον η Γερμανία και η Γαλλία κατανόησαν καλά ότι τα συμβούλια και τα διοικητικά συμβούλια με την ισότητα των φύλων μπορούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η δική μου χώρα, δυστυχώς η Ολλανδία, δεν το κατανόησε και δεν προχώρησε και οι Ολλανδικές επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύονται το, τα, το ταλέντο και την, τις δυνατότητες των γυναικών. Ήδη στο κατόφλι προσλήψεων αποτυγχάνουν οι προσλήψεις των γυναικών. Προτείνει να αναζητηθεί μια λύση η Λουξεμβουριανή Προεδρία στην, στο πάγωμα αυτού του, στην, του ζητήματος στο Συμβούλιο. Πρέπει όμως κατεπηγόντως να υπάρξει δράση, να υπάρξει ένα συμβιβασμός, γιατί η Ολλανδική Προεδρία δεν θα επιτευχθεί αυτό. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιονγκέριους. Για 1,5 λεπτό τώρα ο συνάδελφος Σέινφελντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ιδιαίτερα ευαίσθητο Στη σημερινή κοινωνία κατά τον 21ο αιώνα είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Το ζήτημα είναι ύψης της σημασίας ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα εκεί όπου θα πρέπει να εκπροσωπείται ολόκληρη η κοινωνία. Δεν μιλάμε όμως μόνο για το δημόσιο τομέα, για το δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα έγκυται στον ιδιωτικό κυρίως και έχουμε να κάνουμε με οικονομικές δραστηριότητες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. Μιλάμε για ε, ένα νομικό σύστημα το οποίο ορίζεται από τα κράτη-μέλη που σχετίζεται με την αρχή της αναλογικότητας δυνάμει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Κατανοώ το θέμα των διοικητικών συμβουλίων. Ξέρω ότι το θέμα είναι χρονοβόρο και το θέμα θα μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε το πολιτισμικό μας υπόβαθρο και όχι την νομοθεσία. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Σένφελντ. Για ένα λεπτό η συνάδελφος Νόιχλου παρακαλώ. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, σήμερα συζητάμε αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε ποσόστοση ή όχι. Εγώ λέω κατηγορηματικά, έχουμε εδώ και δεκαετίες μια τέτοια ποσόστοση. Εδώ και δεκαετίες έχουμε μια ανδρική ποσόστοση για τους άνδρες αρκεί να είναι κανείς άνδρας ώστε να μπορέσει να φτάσει σε κάποια αξιώματα. Εμείς οι γυναίκες σκεφτόμαστε αν τα προσόντα μας είναι αρκετά ή όχι. Το επαναλαμβάνω. Εδώ και δεκαετίες έχουμε ανδρική ποσόστοση. Η ανδρική ποσόστοση στη Μάλτα είναι 97,5%. Στο μέσο όρο της Ευρώπης είναι 80% αυτή η ανδρική ποσόστοση. Και να το πω κατηγορηματικά και ρητά, είναι δικαίωμά μας ως, γυναικών, ως γυναίκες που είμαστε και δεν είναι υπερβολικό να απαιτούμε 40% δικαίωμά μας είναι και δεν είναι αυτό κάτι το παράλογο αν ζητούσαμε 60-70% θα μπορούσε να γίνει συζήτηση αν θα ήταν αυτό υπερβολικό ίσως τώρα απαιτούμε αυτό το οποίο μας ανήκει αυτό που έχουν οι άνδρες εδώ και δεκαετίες Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Νόχιλ περνάμε στη διαδικασία Cash τώρα όλοι οι συνάδελφοι ε, μπορούν να ενταχθούν. Αλλά όμως ε, ξεκινάει η συνάδελφος Σούντι, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ισότητα των φίλων και η αρχή, λέει η κυρία Σούλιν, στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ίση ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη δημόσιο, στο δημόσιο βίο και στον ιδιωτικό βίο. Σημαντικότατη υπόθεση. Άσχετα από τη συμμετοχή των γυναικών, στο δημόσιο βίο χρειαζόμαστε αυτό να διασφαλιστεί και στο οικονομικό επίπεδο. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία με την κοινή θέση του Συμβουλίου επί της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012, όπου 40% η ποσόστοση θα καθοριστεί για τις εκπροσώπους των γυναικών, του φίλου δηλαδή που δεν εκπροσωπείται επαρκώς στα Συμβούλια. Πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι η Συμβούλια που όσον αφορά την αναλογία των φύλων είναι ισόρροπα, πιο ισορροπημένα, επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις, διότι οι ικανότητες και οι επιθυμίες και των δύο αμφωτέρων λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σούλιν. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 2012 έχει προταθεί οδηγία ώστε το 40% των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών να αντιστοιχεί στο υποεκπροσωπούμενο φύλλο προκειμένου να βελτιωθεί η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. η νομοθετική πίεση φάνηκε να επηρεάζει τα ποσοστά εκπροσώπηση στα δύο φύλλα αφού τον οκτώβριο του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στο ποσοστό εκπροσώπηση των γυναικών σε εισηγμένε στο χρηματιστήριο εταιρείε σε σχέση με το 2010. Έτσι ήταν 11,9% το 2010 και έφτασε στο 21,2% ωστόσο στι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα ποσοστά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση τη γαλλία τη γερμανία και τη φιλανδία όπου τα ποσοστά ξεπερνούν το. 25%. άλλωστε οι γυναίκε, ειδικά σε περίοδο οικονομική κρίση πλήττονται άμεσα περισσότερο από άλλε ομάδε, και αυτό έχει ήδη φανεί. η μειωμένη απασχόληση των γυναικών είναι εμφανής λοιπόν σε όλου του κλάδου και όχι μόνο στι εισηγμένε εταιρείε. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε κύριε Μαριάς. Κύριε Μαριά, ακολουθεί ο συνάδελφος Γιάκοψιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην ορθή πορεία, στο σωστό δρόμο. Όμως, ο στόχος πόρο απέχει ακόμα από εμάς όταν ήμουν νεότερος εξεπλάγει κάπως από το γεγονός ότι χρειάζονται ποσοστώσεις. Μετά όμως από 25 χρόνια στην πολιτική πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η μόνη οδός, η μόνη οδός προς την επίτευξη της ισότητας των φίλων. Πρέπει να διαρωτηθούμε τι θα έκανε το Κοινοβούλιο, ποια θα ήταν η μορφή του αν δεν θα είχαμε ποσόστοση για τις γυναίκες ιδιαίτερα κάνοντας λόγο για αυτό το θέμα, αυτό ισχύει και στο περιφερειακό επίπεδο για τις τοπικές ε, ε, αρχές ε, και δήμους και κοινότητες. Εξεπλάγει λοιπόν από την αναφορά των ανδρικών λέει ποσοστώσεων. Πρέπει να είμαστε όμως ειλικρινείς και ευθύς στις συζητήσεις μας. Τέτοιες δηλώσεις δεν είναι επικοδομητικού χαρακτήρα νομίζω. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Γιάκοφτσίτσα. Από πλευρά ε, παρεμβάσεων συνάδελφε Έθεριτζ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 40% ποσοστό γυναικών σαν δεσμευτικό κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διοικητικά συμβούλια ανέφερε ο Επίτροπο. Η αδίποτε επανέμβαση σε αυτή την κλίμακα είναι ομή παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά από πλευρά κράτου. Χωρί ελεύθερε αγορέ και επιχειρήσει ελεύθερη αγορά δεν έχει ελεύθερου ανθρώπου. Αυτό που θα πρέπει να βλέπουμε είναι ισότητα ευκαιριών. Όχι ισότητα αποτελέσματος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι σημαντικότατο το ότι οι πολιτικοί και οι καλοπροαίρετες ε, κρατικές αρχές να μην αρχίζουν να αποκλείουν ελευθερίες για να έχουν, πετυχαίνουν αξιέπαινους στόχους. Ελευθερία για τις ευκαιρίες. Είναι το μόνο που έχει σημασία σε, ένα, σε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία. Ευχαριστούμε συνάδελφε Έθριτς. Από ε, παρεμβάσει ο συνάδελφος Πολτσακ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο κύριε Πρόεδρε. Παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά να το σκεφτούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Το πεπρωμένο ή ο Θεός ή η μοίρα αποφασίζει ποια είναι η αναλογία στις κοινωνίες μας και αυτή η αναλογία είναι 51% γυναίκες έναντι 49% των ανδρών. Αυτή είναι η φυσική αναλογία των πραγμάτων. Δεν είμαι κατά του στόχου της ποσόστοσης 40% για τα συμβούλια επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει παρέκκληση από την αναλογία αυτή, την αναλογικότητα, υπάρχει μια φυσική κατάσταση. Μια ελεύθερη αγορά δεν νομίζω ότι είναι ο πιο αποφασιστικός παράγοντας εδώ. Όμως, ας θέσουμε εντάξει τα του οίκου μας. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτυγχάνει την ποσόσωση του 40%. Δείξτε μου στο δημόσιο βίο την ποσόσωση του 40% ή την προσέγγιση της φυσικής αναλογίας 51% των γυναικών, 49% για τους άνδρες. Και τότε θα επιτευχθεί ο στόχος της επιχειρήσης. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Πότσεκα. Και στο τέλος τώρα έχετε εσείς συνάδελφε τον Σας ευχαριστώ για τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους που αγωνίστηκα σε έναν κόσμο που βρίσκεται υπό κυρίαρχο ρόλο των ανδρών και σε αυτούς τους κύκλους εργαστήκαμε και εργαστικά και στο Κοινοβούλιο. Όμως η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτύχει την ισότητα των φύλων. Είμαι φιλελεύθερη και νομίζω ότι οι επιχειρήσεις μπορούν οι ίδιες να ε, επιλέξουν πώς θα πρέπει να εκπροσωπούνται στα συμβούλια οι γυναίκες και οι άνδρες. Πρόκειται και για τα δικαιώματα κυριότητας και ιδιοκτησίας ε, και αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και εμβέλεια. Και θεωρώ επίσης ότι τους λάθος στόχους ε, θέλουμε να υλοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε ίσο χρόνο για τη γονεϊκή μέρημνα, καλή προστασία και για τα θέματα ανατροφής των παιδιών ώστε γυναίκες και άνδρες να συμμετέχουν ίσα, με ίσο τρόπο. Πολλές γυναίκες σήμερα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη σταδιοδρομία τους και να γίνουν νοικοκυρές. Δεν μπορεί όμως να αντέξει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχει νοικοκυρές που θα έχουν εκπαιδευτεί σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πάει χαμένο το ταλέντο τους. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Βίξτρομ. Πιο πριν είπα ότι μπορούν όλοι να παρέμβουν όσοι ζήτησαν τον λόγο. Στη συνέχεια όσοι ζητούν να παρέμβουν δεν μπορούν όμως να καλυφθούν. Ο χρόνος πιέζει. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και εξ ονόματος του Συμβουλίου ο κύριος Υπουργός Σμιτ έχει τον λόγο παρακαλώ. Euh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εδώ και 60 χρόνια περίπου στη συνθήκη της Ρώμης άντρες που δεν ήταν πολύ προχωρημένοι όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών ακόμα συμπεριέλαβαν στη συνθήκη την αρχή της ισότητας των μισθών ανδρών και γυναικών. Εκπληκτικό, διότι τότε η διαφορά, η μισθολογική ανδρών γυναικών ήταν γιγαντιαία. Γιγαντιαία λέγω. Σήμερα ακόμα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι μετά από 60 χρόνια, μετά την σύνταξη της συνθήκης της Ρώμης, υπάρχει διαφορά μεταξύ των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Φανταστείτε, αν δεν είχαμε αυτή τη διάταξη τότε στη συνθήκη της Ρώμης, έχω αμφιβολίες ότι θα ήμασταν εκεί που είμαστε σήμερα, ακόμα και αν η παρούσα κατάσταση ακόμα είναι άκρος ανικανοποιητική. Αυτό που προτείνεται δεν είναι το ευκταίο, διότι το ευκταίο θα ήταν η ισότητα να έχει υλοποιηθεί. Να μην διεξάγεται συζήτηση για την πρόθεση των γυναικών, διότι η κατάσταση θα ήταν κανονική, θα υπήρχαν 60% καμιά φορά 60% γυναίκες αλλού. Ξέρετε η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, θα πρέπει τώρα, τώρα να υπάρξει ένα μέσο, ένα εργαλείο, ούτω ώστε να μην πρέπει να περιμένουμε 70 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα, 90 χρόνια, όπως είπε κάποιος. Εγώ δεν ζήτησα υπομονή. Είπα ότι θα ήταν πολύ να, να ζητήσουμε και υπομονή. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, με ρωτήσατε. Η θέση του Συμβουλίου δεν είναι τόσο διαφορετικές από κάποιες τοποθετήσεις που άκουσα εδώ. Καμιά φορά αναφέρεται επικουρικότητα, καμιά φορά δεν υπάρχει συμφωνία για υποχρεωτικό μέσο. Καμιά φορά μιλάνε για την ελεύθερη επιχείρηση ε, που θα κάνει τη σωστή επιλογή. Υπάρχει ποικιλομορφία στο Συμβούλιο που αντικατοπτρίζει αρκετά καλά την ποικιλία των θέσεων που εκφράστηκαν εδώ. Σας εγγυώμαι λοιπόν ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και λίγο παραπάνω μάλιστα, αλλά η ειδική πλειοψηφία είναι η ειδική πλειοψηφία. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να την πετύχουμε και σίγουρα θα εργαστούμε προς αυτό το σκοπό. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως όλες τις εγγυήσεις γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ Σμιτ είναι γενικά καλό όταν δίνονται υποσχέσεις, αλλά μην υποσχόμαστε